και επίσης το γεγονός οτι ότι κάποια κράτη-μέλη δείχνουν αυτή την περιφρόνηση προς τους υπόλοιπους. Και έτσι αργούμε να πάρουμε τις αποφάσεις και κάνουμε λίγα πράγματα. Πολλοί Ευρωπαίοι να αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, πότε θα κάνουμε κάτι. Πότε θα δράσουμε ενωμένοι, φιλόδοξα και με αλληλεγγύη τώρα που οι Ευρωπαίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Πρέπει τώρα να δράσουμε φιλόδοξα Ευχαριστούμε κύριε Λόπες. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό η κυρία Βίσελερ Λίμα. Το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία όπως το COVID-19 είναι πρώτα να αντιμετωπίσουμε ε, την ασθένεια, να προστατεύσουμε τα θύματα, να προστατεύσουμε τους ασθενείς και τους ε, συγγενείς τους. Και βεβαίω χρειάζονται και αποφάσεις οι οποίες περιορίζουν ελευθερίες. Ε, ε παίρνουμε μέτρα ε, τα οποία είναι έκτακτη ανάγκη. Όμω θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι το κράτο δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα θα προστατεύονται. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε, να παρακολουθήσει η Κομισιόν σαφώ τα εξαιρετικά μέτρα που παίρνουν οι εθνικέ κυβερνήσει και να παρέμβει εφόσον υπάρχουν παρεκκλήσει και ολισθήματα. Θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει το ρόλο του το Κοινοβούλιο ω νομοθέτη και ω ελεγκτή. Αυτή η κρίση δείχνει πόσο εξαρτώμεθα ε, από άλλες ε, χώρες σε εξοπλισμό σε είδη πρώτης ανάγκης. Όταν μιλάμε για Τώρα μιλάμε για υλικό ιατρικό, αλλά αυτό μπορεί να ισχύσει και για διατροφή στο μέλλον. Τι περιθώριο λιγμών έχει η Κομισιόν απέναντι στην Κίνα όταν εξαρτάται από ε, τις ε, εισαγωγές μασκών η Κίνα, παραδείγματο χάρη, ε, δεν δέχεται να μπει η Ταϊβάν στον ΠΟΗ. Εμεί δεν αντιδρούμε σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε πιο ισχυροί, να προστατεύσουμε τι υποδομέ μα, τι βιομηχανίε μα και στη διεθνή πολιτική σκηνή να μπορούμε να υπακούσουμε τις πεπιθήσεις μας και να είμαστε ε, αλληλέγγυοι προς τους πληθυσμούς που εκτίθενται περισσότερο ανά τον κόσμο. Ευχαριστούμε κυρία Βίσλερ Λίμα. Για ένα μισή λεπτό ο Σπίτσουλα. Πίτσουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όποιος ε, θέλει βρίσκει τον τρόπο. Αυτή η δυστυχή συγκυρία θα πρέπει να μας εμπνεύσει για το μέλλον, για παράδειγμα το πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Φαίνεται τόσο ασήμαντο το να μαζέψεις το 1 ή το 1,7%. Πρόκειται για τη χειρότερη κρίση που μας έχει πλήξει μετά από τη δεκαετία του 1930. Όσον αφορά τα ταμεία συνοχής θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να μετριάσουμε τις συνέπειες της κρίσης τα ταμεία συνοχής, τα κονδύλια ταμείου συνοχή είναι αυτά που θα τελευταία θα πρέπει να περικοπούν στον μελλοντικό προπολογισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό μας για να αγοράσουμε προστατευτικό εξοπλισμό και να υποστηρίξουμε τα συστήματα υγειονομική περίθαλψης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα fake news και να μην ξεχνάμε να προσέχουμε να μην είναι κακή ποιότητα, ε, οι μάσκες και ο προστατευτικό εξοπλισμό σε όλο τον κόσμο. Επίση, τα κονδύλια για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί σε αυτέ τι αγροτικέ περιοχέ, είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή την κρίση. Οι συνέπειε αυτή τη κρίση θα πρέπει να μετριαστούν με τεράστια ε, ποσά δημόσια αλλά αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν με διαφάνεια και υπεύθυνα σε όλα τα επίπεδα. Για να κλείσω, θέλω να υποστηρίξω αυτή την πολιτική συμφωνία. Αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα, αλλά η πολιτική μας συμφωνία είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή για να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτσουλα. Ακολουθεί για μισή λεπτό ο κύριος Κάζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα κοινό εχθρό ένα εχθρό που δεν ξέρουμε από πού ήρθε και πού πάει. Η Ευρώπη ντρέπεται. Σε τέτοιε εποχέ κρίση είναι σημαντικό να συντονίζουμε τη δράση μα και αυτή είναι ένα αποφασιστική. Καλωσορίζω αυτό το ψήφισμα που θα μα βοηθήσει να σώσουμε ζωέ και μέσα διαβίωση. Υπάρχει περίπτωση ότι η διαφωνία να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερες ζημιές. Ε, είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να προχωρήσουν βάσει αυτής της πρότασης αλλά να πάνε και πιο πέρα. Πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά των οικονομιών μας. Να υπάρχει πρόσβαση για να τις υποστηρίξουμε γρήγορα τώρα και στο επόμενο ε, χρηματοπιστωτικό διάστημα. Και επίσης να ενισχύσουμε τα υγειονομικά μας συστήματα, το MFF και το ESF Plus το οποίο εγώ είμαι αρμόδιο, είναι σημαντικό εργαλείο από αυτή την άποψη. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η χρηματοδότηση να συνεχίσει να ρέει. Και εμεί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλιστεί ότι τα νέα κονδύλια θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν του χρόνου. Ταυτόχρονα πρέπει να προετοιμάσει μέτρα έκτακτη ανάγκη η για όσου θα έχουν ανάγκη. Κύριε Πρόεδρε, οι πολίτε μα εξαρτώνται από εμά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι περιστάσει. Δεν πρέπει να του απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάζα. Τώρα η κυρία Ντυπών για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν ε, είπε ε, για τη θητεία της μια ένωση που προσπαθεί για περισσότερα. Ε, έδρασε γρήγορα και σωστά η Ευρώπη. Στην Ολομέλεια του Μαρτίου ψηφίσαμε το πρώτο πακέτο με μέσα ε, διάσωσης για του πολίτε, για τι επιχειρήσει, με την απαραίτητη ευελιξία. Εμεί αυτή τη βδομάδα ψηφίζουμε και συμφωνούμε το επόμενο πακέτο με νέα μέτρα για την άρση των ε, ε, περιορισμών που υπάρχουν από τη γραφειοκρατία αλλά ορισμένα κράτη-μέλη είναι πράγματι έδρασαν ταχύτερα. Σε ορισμένε περιπτώσει είχαν δίκιο και παρόλα αυτά αυτό είχε ω αποτέλεσμα να γίνουν και κάποια μη αναγκαίε προσπάθειε και να γίνουν και κάποιε μη αναγκαίε εντάσει μεταξύ κρατών μελών. Κύριε Επιτροπέ, μια η Ευρώπη που προσπαθεί για περισσότερα εξακολουθεί να ισχύει και είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ. Όλοι αντιμετωπίζουμε αβεβαιότητα, άγχος, δεν υπάρχει κάτι, κάποιο προηγούμενο που να μας καθοδηγεί. Είναι ήδη τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με τον ιό που προκαλεί οδύνη στους πολίτες μας. Είμαστε όλοι κοντά στον, στους άλλους και αισθανόμαστε τον πόνο των γειτόνων μας, των άλλων Ευρωπαίων πολιτών που ε, πλήττονται περισσότερο. Καθώ ζητάμε από του πολιτέ μα να παραμένουν σπίτι, να κρατούν αποστάσει από του άλλου, οι δικέ του προσπάθειε θα πρέπει να καθοδηγούν εμά. Καθώ προσπαθούμε να μετριάσουμε τι συνέπειε τη κρίση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, να διαπραγματεύσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα. Ε, στηριχθείτε πάνω μα για να καταπολεμήσουμε με ευρωπαϊκέ απαντήσει τον ιό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο όλοι και όπω έχει το σλόγγαν του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είναι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί καλύτερα. Ευχαριστούμε κύριε Ντυπών. Τέλος ο κύριος Επίτροπος, κύριος Σεφτσοβίτς. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν εδώ την περασμένη φορά και μιλήσαμε για τους ήρωες του σήμερα, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες, αυτούς που εργάζονται στα καταστήματα, την αστυνομία, τους εθελοντές που βοηθούν τους ηλικιωμένους, τους πιο ευάλωτους. Σήμερα Όπω πολύ σωστά είπε και η κυρία Ντυπό, θα πρέπει να εκφράσουμε την εκτίμησή προ προς συμπολίτε μας, οι οποίοι μας αποδεικνύουν ότι είναι εξαιρετικά υπεύθυνοι, σεβόμενοι τους κανόνες, μένοντας σπίτι, σεβόμενοι την κοινωνική απόσταση, που είναι δύσκολο όταν κάποιο εργάζεται στο σπίτι του, έχει παιδιά. Και βεβαίως αυτή η συζήτηση απέδειξε ότι η Ευρώπη έρχεται να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Είχαμε πολλά παραδείγματα όπως ε, οι άνθρωποι αλλά και τα κρατημέλη βοηθούν ο ένας τον άλλον, πώς μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση και πώς προετοιμαζόμαστε για την ε, οικονομική κρίση που ακολουθεί. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω, σας ευχαριστήσω όλους όλα τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενέργειά σας, για την υπομονή σας, αλλά και διότι εκφράσατε, αυτά που νιώθουν οι πολίτες τους οποίους εκπροσωπείτε. Η κρίση του COVID ε, περιγράφεται από κάποιους ως ε, ένα δραματικός επιταχυντής, επιταχυντής και καλού. Ε, βλέπουμε ο ηρωισμός, η ευθύνη πολλών ανθρώπων, η υπευθυνότητα που βοηθούν στο να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η κοινωνία παρά την κρίση. Είδαμε πως η λήψη των αποφάσεων ε, επιταχύνθηκε. Συμφωνώ με τον κύριο Μουρεσάν. Πραγματικά σε λίγε εβδομάδε, εβδομάδες, 4-5 εβδομάδε κάναμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε ε, τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης από ό,τι κάναμε ε, μέσα σε 4 χρόνια ε, στην προηγούμενη χρηματοοικονομική κρίση. Για να, είμαι όμως, για να είμαστε όμω ειλικρινεί, ε, υπάρχει και ένα αρνητικό στοιχείο. Fake news, ψευδείς ειδήσει, επικίνδυνος λαϊκισμός, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία μας δοκιμάζονται. Το είπε και ο κύριος Λάμπερς νωρίτερα και θέλω να πω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά επαγρυπνούμε σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη και είμαστε σε στενή επαφή και με την Ουγγαρία και με την Πολωνία και αναλύουμε βεβαίω όλες τις ψευδείς ειδήσει, όλο, όλο αυτόν τον αρνητισμό ε, τον οποίο διαχέεται στα κοινωνικά μέσα δικτύωση ζητούμε την ελαχιστοποίηση αυτών των, των ε, ε, φαινομένων και μα ακούνε ο κ. Κοντάλες Πόνς, η κυρία Γκαρσία Πέρεθ, ο κύριος Τσόλος πολύ σωστά είπαν ότι το μέλλον της Ευρώπης αποφασίζεται τώρα και αυτό που χρειαζόμαστε ε, μια Ευρώπη πιο δημοκρατική, πιο πατριωτική, πιο ισχυρή και θέλω να σας, ευχαριστήσω όλους που εκφράσατε σαφώς τις απόψεις σας για το πόσο χρειαζόμαστε μαζικές οικονομικές επενδύσεις. Ελπίζω σήμερα να υποστηρίξετε το πακέτο το οποίο έχει ως σκοπό να προσφέρει άμεσα μέτρα ενίσχυσης. Αλλά θα πρέπει βεβαίως να επενδύσουμε μαζικά και στην ανάκαμψη, να διαφυλάξουμε ε, τις θέσεις εργασίας, να προστατεύσουμε ε, την ε, οικονομία μας ε, σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Marshall για το μέλλον της Ευρώπης, αλληλέγγυο, βιώσιμο, καθαρό, ψηφιακό και βεβαίως πιο ανθεκτικό όπως είπαν πολλοί από εσά. Μόνο έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού το μέλλον μας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες της νέας αγοράς, να επωφεληθούμε από την πράσινη επανάσταση αλλά και την ψηφιακή επανάσταση και να μάθουμε και από αυτή την κρίση δημιουργώντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα μια πιο ισχυρή Ευρώπη θα θυμάστε ότι στο παρελθόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές και διάφορες εξαρτήσεις ο λόγος για την εξάρτηση αυτή ε, οι εξαρτήσει αυτή μα δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε στρατηγικοί. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να παράγουμε εμεί οι ίδιοι στην Ευρώπη. Δημιουργούμε τώρα αποθήκε ε, ε, ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού. Θα πρέπει όμως να μην εξαρτώμεθα μόνο από μία χώρα ή από μία εταιρεία. Επίσης θα πρέπει αφού κάνουμε μια σωστή ανάλυση να αποφασίσουμε τι χρειάζεται να παράγουμε εδώ στην Ευρώπη για να είμαστε βέβαιοι ότι όταν θα το χρειαστούμε θα το έχουμε. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι όλοι όσοι είπαν ότι χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη, μια πιο στρατηγική, μια πιο ενωμένη ε, προσέγγιση ε, είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να χρηματοδοτήσουμε αυτή την προσπάθεια. Χρειαζόμαστε ισχυρό ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και διαφορετικό πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει αυτό το προπολογισμό να μπορέσουμε να το φορτώσουμε οικονομικά στο πρώτο κομμάτι τη επταετία. Ε, να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στου τομεί εκείνου όπου χρειάζεται βοήθεια άμεσα, που χρειάζεται βοήθεια άμεσα, να μπορέσουμε να προλάβουμε μελλοντικέ κρίσει και να μπορέσουμε πραγματικά να ανακάμψουμε και στον τομέα της νέας οικονομίας, να δώσουμε μια μάχη και για θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας, όπως είπαν πολλοί από εσά, το είπε ο κ. Μποτεγκά, το είπε, η κυρία Ντελάγκη και πραγματικά ε, θέλω να είμαι εξαιρετικά ανοιχτό απέναντί σας. Ε, πραγματικά εξαρτώμεθα από την υποστήριξή σας για να έχουμε φιλόδοξε σύγχρονες, ε, πολιετές ε, δημοσιονομικές προοπτικές που θα μας βοηθήσουν να, προσ... να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, να εξελονίσουμε την Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε ε, τον οικονομικό αντίκτυπο τον οποίο όλοι περιμένουμε μετά από αυτή την κρίση. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο θέμα του προστατευτικού υλικού των μασκών. Θέλω εδώ να σας διασφαλίσω ότι εργαζόμαστε 24 ώρες 24 ώρο. Οι συνάδελφοι, η Στέγια Κυριακίδη, ο Τιερή Μπρετό, άλλοι επίτροποι, εργαζόμαστε σκληρά και πολύ σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα αυτής της κοινή προμήθειας που θα εξασφαλίσει ότι οι γιατροί μας, οι νοσοκόμες μας, οι πολίτες μας θα έχουν ό,τι χρειάζεται ε, για να μπορέσουν να εργαστούν. Επίσης θέλω να πραγματικά να συγχαρώ τις ευρωπαϊκές εταιρείες που μετατρέπουν την παραγωγή τους για να μπορέσουν να παράξουν μάσκες ή απολυμαντικά ε, τζελ ή παράγουν πλέον και αναπνευστήρες που χρειάζομαστε τόσο πολύ στα νοσοκομεία μας και πραγματικά πιστεύω ότι σε λίγους μήνες αυτή η ισχυρή ε, ε, δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ε, θα φέρει πολύ, πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έγινε αναφορά ε, στο θέμα των ηλικιωμένων και των πιο ευάλωτων. Η μητέρα μου ε, και η πεθερά μου βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στη Σλοβακία. Έχουμε τροποποιήσει το σχετικό ταμείο για τους πιο ευάλωτους, τους πιο φτωχούς, να δούμε αν αρκεί αυτή η μετατροπή, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ε, για να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται από τη μεγαλύτερη βοήθεια. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αντιδράσω σε δύο πολύ σημαντικά σχόλια. Το ένα του κύριου Γκασπαρή, ο οποίος ανέφερε το ζήτημα ε, της ε, εφαρμογής ιχνηλάτησης του ιού. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή εφαρμογή με την καλύτερη πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη. Μια εφαρμογή που θα εχνηλατεί τον ιό, όχι ανθρώπους. Θα σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα είναι θελοντική για όσους θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν, θα είναι ανώνυμη και θα λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να σας ενημερώνει μέσω ενός SMS ότι ενδεχομένως να έχετε εκτεθεί στον ιό και θα πρέπει να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα. ο κύριος Φερχόπστα, η κυρία Σπυράκη, ο κύριος Λαρουτουρίου, η κυρία Σίλβαντε Περέιρα έθεσαν το ζήτημα του σχέδιου ανάκαμψη στα πλαίσια του πολιτισμού πολιτισμικού πλαισίου. Προσπαθούμε λοιπόν και εμεί να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα εργασιών τη Κομισιόν, το οποίο θέλουμε να σα υποβάλουμε πριν το τέλο του μήνα. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα μέτρα, όπω είπε και η κυρία Φόντερ Λάιεν, κατέθεσαν εφικτό σε ένα πολύ μικρό διάστημα να κινητοποιήσουμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Συμφωνώ μαζί σα ότι χρειαζόμαστε περισσότερα. Και πιστεύω ότι με τη δική σα υποστήριξη μπορούμε να έχουμε καλέ πολιτέ δημοσιονομικέ προ... προοπτικέ. Ξέρουμε όμω ότι χρειάζεται και διπλωματία, διότι οι αποφάσει για το ΠΔΠ παίρνεται ομόφωνα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε και εργαζόμαστε εντατικά. Μιλούμε με του αρχικού κανόνε κυβερνήσεων στην πρόταση που θα υποβάλουμε να είναι αρκετά φιλόδοξη, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσει να τύχει τη υποστήριξη όλων των κρατών μελών τη Ένωση, διότι αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μάθουμε το παρελθόν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευση, να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες πολιτικές μας που, φέρουν, που, παρέχουν καλές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Και όλα αυτά πιστεύω θα αποτυπωθούν στις μελλοντικέ μας προτάσεις. Τελειώνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις σας και για την υποστήριξη που εκφράσατε και όλες αυτές τις περασμένες δύσκολες εβδομάδες ελπίζω με την υποστήριξή σας να δημιουργήσουμε μια νέα, να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη που θα προκύψει από αυτή τη δραματική κρίση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επιτρόπε, κύριε Σεφτσοβίτς. Ο κύριος ε, Μισελ ε, μου ζήτησε να σας μεταφέρω τη συγγνώμη του, διότι χρειάστηκε να φύγει νωρίτερα παρακολουθούν οι συνεργάτες του φυσικά τη συζήτηση και θα εκφράσουν τις ε, απόψεις τους για τα όσα είπαν οι ευρωβουλευτές. Συνεχίζουμε στη μία και μισή μέχρι εκείνη την ώρα. Ε, βρείτε κάτι να φάτε ή φάτε αυτά που φέρατε. Καλή σας όρεξη. Τι ακόπτεται η συνεδρίαση.